Με χαρά λοιπόν θα συνεργαστώ μαζί σας. Η κατάσταση καταλαβαίνω ότι για σας δεν είναι καθόλου εύκολη και ξέρω πως η συνάδελφος την οποία αποχαιρετήσαμε έβαλε πολύ ψηλά τον πύχη. Είμαι όμως πεπισμένος πως η συνεργασία μας θα φέρει πολύ θετικά αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ για λοιπόν να μιλήσουμε και για το θέμα της Γερμηνίας. Έχουμε 21 γλώσσες εδώ και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Νταντά, ο οποίος θα κάνει μια εισαγωγή στο σημείο 3 της ημερήσιας διάταξης, δηλαδή θα μιλήσουμε για το θέμα της ψηφοφορίας και δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάποια εισαγωγή, νομίζω ότι απευθείας μπορείτε να τα πείτε εσείς. Κύριε Πρόεδρε, να σας πω δύο λόγια καταρχήν. Νομίζω ότι όλοι μας ενημερωθήκαμε για ε, το κείμενο το οποίο μας έστειλε ε, η γραμματεία έχει ξεχαστεί κάτι από το κείμενο για τις ψηφοφορίες. Στη σελίδα 15, τουλάχιστον στο δικό μου κατάλογο ψηφοφοριών, είναι στη σελίδα 15 και πρέπει να σας πω στο κεφάλαιο 2, παράγραφος 7, υπό 3, μεταξύ της τροπολογίας 324 και της 61 θα πρέπει να προσθέσουμε την 156 η οποία ξεχάστηκε. Θα ήθελα επίσης να σας πω πως μετά την συνεδρίαση των σκιώδων εισηγητών κάναμε μία συζήτηση για την κλωνοποίηση και η πλειοψηφία των ομάδων εκφράστηκαν με τρόπο που με οδήγησαν στο να μην στηρίξω τις τροπολογίες σχετικές με την κλωνοποίηση στο κείμενο αυτό και να ζητήσω στην αρχή του τριμερούς διαλόγου να κάνω μια δήλωση το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να έχουμε συγκεκριμένο κείμενο για τεχνολογία κλωνοποίησης και την ε, προσαρμοσμένη σε αυτή την τεχνολογία ε, νομοθεσία. Αυτά γιατί θεώρησα πως είμαι ανίκανος να κρίνω μια νομοθεσία ε, περί τεχνολογίας την οποία δεν κατέχω, δεν ελέγχω και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει ένα κείμενο το οποίο θα καλύψει τα τεχνολογικά θέματα στα οποία θα νομοθετήσουμε ε, ξέρω πως υπάρχει μεγάλη πλειοψηφία ε, γιατί έχουμε πει πως δεν θα πρέπει να γίνει εμπορική εκμελα, εκμετάλλευση των προϊόντων κλωνοποίησης νομίζω ότι έχουμε συμφωνήσει οι περισσότεροι αλλά δυστυχώς δεν έχω ακόμα κάποιο κείμενο να προτείνω γιατί τρέχει ο τριμέρης διάλογος Εκτός μικροφόνου Σας ευχαριστούμε πολύ. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Ας περάσουμε λοιπόν κατευθείαν στην ψηφοφορία. Δεν έχω την κάρτα μου μαζί μου. Αυτό ήθελα να σας πω απλώς. Ωραία, το λαμβάνουμε υπόψη. Να σας ζητήσω κάτι μόνο στην αρχή. μπορούσατε να εξετάσετε το ακόλουθο. Αν δούμε ότι οι περισσότεροι είναι υπέρ, αν έχουμε μία πλειοψηφία, να μην σας ρωτάω αναγκαστικά αν είμαστε υπέρ κατά αποχές, αν δω ότι οι περισσότερες σηκώνται τα χέρια σας, ε, ότι έχουμε μια πλειοψηφία εξ αρχής, δεν υπάρχει λόγος να λέω όλο αυτό υπέρ, κατά, αποχές κτλ. Θα εξοικονομήσουμε χρόνο κατά αυτόν τον τρόπο. Θα σας λέω απλώς, λοιπόν, θα ρωτάω απλώς στην αρχή ποιο είναι υπέρ, χωρίς να σας ρωτάω στη συνέχεια ποιο είναι κατά ή ποιο απέχει. Πολύ ωραία. Λοιπόν, NV υπαριθμόν 8 πρώτη τροπολογία που ψηφίζουμε. Να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε 157 τροπολογίες από τον εισηγητή και συνολικά 346 τροπολογίες για το κείμενο αυτό και 12 συμβαστικές τροπολογίες. Τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Άρτη ψηφοφορία ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρες. Εγκρίνεται. 32 υπέρ και 5 κατά. 186 υπέρ παρακαλώ. Ευχαριστώ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 16. Υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 17. Υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία Α. ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται η συμβαστική τροπολογία Α. Περνάμε στην τροπολογία 192 υπέρ παρακαλώ. 192 κατά απορρίπτεται 193 υπέρ κατά απορρίπτεται τροπολογία 194 υπέρ παρακαλώ κατά απορρίπτεται συμβαστική τροπολογία β άρτη ψηφοφορία ηλεκτρονικά περες κρινεται Κρίνεται. NV11 υπέρ κατά απορρίπτεται. Τροπολογία 107 υπέρ κατά Απορρίπτεται. Περνάμε στη συμβαστική τροπολογία C. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά, άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 21 του εισηγητή υπέρ παρακαλώ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 203 υπέρ εγκρίνεται. Τροπολογία 204 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 205 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 206 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 22 του εισηγητή και 13 της ένδυ υπέρ, εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 23, η οποία είναι πολύ σημαντική και θα ψηφίσουμε γι' αυτό ηλεκτρονικά άρτη ψηφοφορία για την τροπολογία 23. Κάνει με την κλωνοποίηση η τροπολογία αυτή, πέρας. Το ήξερα, μα το ήξερα. Είναι πολύ βασική όμως τροπολογία αυτή, ιδιαίτερα θεμελιώδης, γι' αυτό το λόγο ήθελα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά και αυτό θα κάνουμε και σε δύο κόμμα τροπολογίες. Μολονότι βέβαια ήξερα ότι το αποτέλεσμα θα ήταν αυτό που είδαμε, εγκρίνεται προφανώς. 14 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 15 υπέρ, εγκρίνεται. Τροπολογία 209 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 24, ταυτόση με τη 210 και τη 16 Τη ΣΕΝΒΗ, υπέρ παρακαλώ, εγκρίνονται. 25 υπέρ, εγκρίνεται. 26 υπέρ, εγκρίνεται. Τροπολογία 211. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία αυτή. 211. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 212. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά και για αυτή την τροπολογία. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Κύριε Χάουσλινγκ, 2.13 του κυρίου Χάουσλινγκ εγκρίνεται, 2.14. Πολύ σημαντική τροπολογία αυτή. Ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για τροπολογία 214. Πέρας. Απορρίπτεται. Περνάμε στην τροπολογία 215. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Απορρίπτεται. 216. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 27. Υπέρ. Συμβαστική τροπολογία D. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 31. Υπέρ παρακαλώ. Ευχαριστώ. Συμβαστική τροπολογία E. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην 227 υπέρ παρακαλώ του κυρίου Χάουσλεν η τροπολογία αυτή κατά απορρίπτεται. Τροπολογία 36 υπέρ μάλλον δεν την ψηφίζουμε 36 36 του εισηγητή υπέρ παρακαλώ εγκρίνεται 228 υπέρ κατά απορρίπτεται Περνάμε στην συμβαστική τροπολογία F, άρχεται ψηφοφορία, πέρας. Ευχαριστώ, εγκρίνεται. 43. Υπέρ παρακαλώ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 45. Υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 46 υπέρ. Εγκρίνεται. ...232 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Περνάμε στην συμβαστική τροπολογία G, άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 49. Του εισηγητή υπέρ παρακαλώ. Εγκρίνεται. 240 Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Εγκρίνεται. 241. Ευχαριστώ. Απολογία 50. Υπέρ παρακαλώ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 51. Του εισηγητή υπέρ. Εγκρίνεται. Προπολογία 52 υπέρ. Εγκρίνεται. 53 υπέρ. Εγκρίνεται. 54 υπέρ παρακαλώ. Εγκρίνεται. 55 υπέρ παρακαλώ. Εγκρίνεται. 56 υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 57 υπέρ παρακαλώ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 58 και 249 υπέρ εγκρίνονται. Συμβαστική τροπολογία H ψηφίζουμε ηλεκτρονικά άρθρη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Και περνάμε στην τροπολογία 251 υπέρ παρακαλώ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 60 υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 61 υπέρ. Εγκρίνεται. 252 υπέρ. Εγκρίνεται. 62 υπέρ εγκρίνεται. 254 υπέρ παρακαλώ εγκρίνεται. 63 υπέρ. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 254. Άρτη ψηφοφορία. Υπέρ. Κατά. Ψηφίζουμε την τροπολογία 254. Υπέρ παρακαλώ. Ας ελέγξουμε μάλλον ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 254. Άρτη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 63 υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 255 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 250, μάλλον. Πρώτα θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 255 άρτη ψηφοφορία. Πέρας. κρίνεται, συγγνώμη. Περνάμε στην τροπολογία 256, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 257. Μάλλον 64 διορθώνει ο πρόεδρος. Ψηφίζουμε τροπολογία 64. Υπέρ παρακαλώ. Κύριο Σάγνιο Κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχει αγγλική μετάφραση για τη 257, για τη 257 δεν ξέρω τι ψηφίσαμε, δεν ήξερα γιατί ψηφίζαμε και δεν μπόρεσα να ψηφίσω. Αλλά από ό,τι φάνηκε και κάποιοι άλλοι δεν ψήφισαν τελικά. Μα δεν, δεν ψηφίσαμε την 257, πίπτη γιατί εγκρίναμε τη 256, γι' αυτό δεν την ψηφίσαμε. Ναι. Καταπίπτει όπως σας είπα. Λοιπόν, τροπολογία 64 υπέρ παρακαλώ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 65 υπέρ. Εγκρίνεται. Περνάμε στην συμβαστική τροπολογία I. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 68 του εισηγητή. Υπέρ παρακαλώ. Ευχαριστώ. Εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 69. Υπέρ παρακαλώ. Εγκρίνεται. Φτάσαμε στην συμβαστική τροπολογία J, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Και περνάμε στην τροπολογία 71 και 32 της ΕΜΒ, υπέρ παρακαλώ, εγκρίνονται. Τροπολογία 33. Υπέρ. Εγκρίν. Ευχαριστώ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 33. Άρθη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με μικρή πλειοψηφία, αλλά εγκρίνεται. Τροπολογία 72 υπέρ, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία K, άρχιτη ψηφοφορία, πέρας, εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 278, υπέρ παρακαλώ, κατά, Απορρίπτεται. Τροπολογία 74 υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 279 και 75 μαζί. Υπέρ παρακαλώ. Εγκρίνονται. 76 υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 77 υπέρ. Εγκρίνεται. 78 υπέρ. Εγκρίνεται. 79 υπέρ εγκρίνεται. Τροπολογία 80 υπέρ εγκρίνεται. Τροπολογία 281 υπέρ παρακαλώ κατά απορρίπτεται. Τροπολογία 81 του εισηγητή υπέρ εγκρίνεται. Τροπολογία 82 υπέρ, εγκρίνεται. Τροπολογία 36, υπέρ, εγκρίνεται. Τροπολογία 282, υπέρ, εγκρίνεται. 283, 284, με συγχωρείτε, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 84 του εισηγητή υπέρ κα, εγκρίνεται λοιπόν 85 του εισηγητή υπέρ εγκρίνεται 285 υπέρ 85 εγκρίνεται άρα λοιπόν η 285 καταπίπτει 86 υπέρ της 86 εγκρίνεται 87 υπέρ. Εγκρίνεται. 88 υπέρ. Εγκρίνεται. 89 υπέρ. Εγκρίνεται. 287 υπέρ. Απορρίπτεται. 288 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 90 υπέρ. Εγκρίνεται. 91 υπέρ εγκρίνεται 92 του εισηγητή υπέρ εγκρίνεται 289 υπέρ εγκρίνεται 2.92 υπέρ κατά απορρίπτεται. Επόμενη τροπολογία 2.93 υπέρ κατά απορρίπτεται 2 Όχι. Μπορούμε να περάσουμε στην 2.96. Η 2.96 υπέρ. Εγκρίνεται. 2.97 υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 93 υπέρ εγκρίνεται 301 υπέρ κατά απορρίπτεται 302 υπέρ 302 υπέρ εγκρίνεται η 95 του εισηγητή υπέρ εγκρίνεται 303 υπέρ 303 υπέρ εγκρίνεται Μπορούμε να περάσουμε λοιπόν στην τροπολογία υπαριθμών 104. 104 υπέρ. Με συγχωρείτε, διορθώνει προς 102. 102. 1, 102 του εισηγητή. Υπέρ. Εγκρίνεται. Και η επόμενη είναι η 104 τώρα. 104 υπέρ εγκρίνεται 105 υπέρ εγκρίνεται 106, 106 με συγχωρείτε υπέρ εγκρίνεται 107 υπέρ εγκρίνεται η 39 έμβη υπέρ εγκρίνεται 108 του εισηγητή υπέρ εγκρίνεται 109 εισηγητή υπέρ εγκρίνεται 110 του εισηγητή υπέρ εγκρίνεται η 40 έμβη υπέρ εγκρίνεται 111 υπέρ εγκρίνεται 112 υπέρ εγκρίνεται 113 υπέρ εγκρίνεται. 114 υπέρ. Ευχαριστώ πολύ. Εγκρίνεται. 115 υπέρ. Εγκρίνεται. 305 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 116 υπέρ. Εγκρίνεται. 306 υπέρ, κατά. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία για την 306 ηλεκτρονικά. Απορρίπτεται. Περνάμε λοιπόν στην 117 υπέρ Περνάμε λοιπόν τώρα στην τροπολογία 41. 41. Ένβη, υπέρ. Στην προηγούμενη ήμασταν 22-22, άρα απορρίπεται. Λοιπόν, περνάμε στο επόμενο που είναι η 41, υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 118, υπέρ. Εγκρίνεται. 119, υπέρ. Εγκρίνεται. 307, υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 120, υπέρ εγκρίνεται 121 υπέρ εγκρίνεται 308 υπέρ κατά απορρίπτεται για να ψηφίσουμε λοιπόν από την 123 με την 134 έχουμε τροπολογίες, μια σειρά τροπολογιών του εισηγητή. Μπορούμε λοιπόν αυτές όλες μαζί να τις ψηφίσουμε με μιας από το 123 μέχρι το 134. Υπέρ. Ευχαριστώ πολύ. Εγκρίθηκαν. Τροπολογία 135 του εισηγητή υπέρ. Εγκρίνεται. 136 υπέρ. 136 υπέρ. Εγκρίνεται. 312, 313, 137 υπέρ. Εγκρίνεται. Μαζί και οι τρεις. 138 υπέρ. 138 υπέρ. Εγκρίνεται. 139 υπέρ. Εγκρίνεται. 43 έμβη υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 141 και 44 υπέρ εγκρίνεται. Περνάμε στο L. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για τη συμβεστική πρόταση L. Άρχεται. Λίγη. Εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην 45 υπέρ. Εγκρίνεται. 315 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 316. Που είναι παρόμοια με τη 46 υπέρ. Εγκρίνεται. 144. 144 υπέρ Υπέρ 144. Ευχαριστώ, εγκρίνεται. 140. Μισό λεπτό. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 48. Έμβη, υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 301 υπέρ 310 με συγχωρείτε 146 που είναι με τη 49 υπέρ εγκρίνεται 319 υπέρ υπέρ 319 υπέρ κατά ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 319 Άρχεται. Λίγη. Ευχαριστώ πολύ. 320 υπέρ. Εγκρίνεται. 321 υπέρ. Εγκρίνεται. 147 υπέρ. Εγκρίνεται. 322. Υπέρ. Υπέρ. 322. Κατά. Απορρίπτεται. 148 που είναι 51 έμβη. Υπέρ. Εγκρίνεται. 149, 53 έμβη. Υπέρ. Εγκρίνεται. 150, 54 έμβη. Υπέρ. Εγκρίνεται. 151 και 55 υπέρ Εγκρίνεται. Τρακόσια υπέρ κατά απορρίπτεται. Θα ελέγξουμε λοιπόν ηλεκτρονικά την 323. Άρχεται. Otwieram głosowanie na poprawkę 323. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Α, εσείς. Ναι, εγκρίνετε τότε. Περνάμε στην τροπολογία 154. Μπράβο σας, εργατικότατοι είστε. 154 λοιπόν και 57 ένβη. Υπέρ εγκρίνεται. 1, 55 και 57 υπέρ. Ευχαριστώ, εγκρίνεται. 3,24 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Μία πρόσθετη τροπολογία την οποία ανέφερε ο κύριος Νταντέν 156 324 κύριε Πρόεδρε μπορούμε να την ελέγξουμε ηλεκτρονικά μετά από έτοιμο του κυρίου Άγνιου ψηφίζουμε ξανά την 324 άρχεται η ψηφοφορία Πέρας Σας ευχαριστώ. Περνάμε λοιπόν στην τροπολογία του κυρίου Νταντάν ή 156. Ποιος είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Εγκρίνεται. 325. Υπέρ. Εγκρίνεται. 326. Υπέρ. Κατά. Η 325 εγκρίνεται και η 326 απορρίπτεται. 327. Ποιος είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Εγκρίνεται. 328. Υπέρ. Εγκρίνεται. 329. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την 329. Άρχεται η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Σωστά. Πράγματι, απορρίπτεται. 330. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 331. Υπέρ. Εγκρίνεται. 332. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 333. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 334. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 335. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 338. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 67. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 339. Υπέρ. Εγκρίνεται. 157. Όχι, ηλεκτρονική επαλήθευση για την 339 άρχεται η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 157 υπέρ. Εγκρίνεται. 341 επί υπέρ κατά. Απορρίπτεται. 342 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 343. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 344. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 158 από τον κύριο Ντόρφμαν. Υπέρ, εγκρίνεται. 159. Υπέρ, εγκρίνεται. 1. Ένβη. Του εισηγητή, υπέρ, εγκρίνεται. 160 υπέρ κατά απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ εγκρίνεται. 3 υπέρ εγκρίνεται. 162 από τον κύριο Άγνιου υπέρ κατά απορρίπτεται. 163 του κυρίου Ντόρφμαν. Υπέρ. Ευχαριστώ. Εγκρίνεται. 164 υπέρ. Εγκρίνεται. 165 υπέρ. Εγκρίνεται. 3 του εισηγητή υπέρ. Εγκρίνεται. 167 υπέρ κατά απορρίπτεται 168 υπέρ εγκρίνεται 4 του εισηγητή υπέρ εγκρίνεται 5 του εισηγητή υπέρ εγκρίνεται 169 του κυρίου Μπούντα υπέρ εγκρίνεται. 7 του εισηγητή και 5 ένβη υπέρ εγκρίνεται. 8 του εισηγητή υπέρ εγκρίνεται. 6 ένβη υπέρ εγκρίνεται. 170 υπέρ εγκρίνεται. 9 υπέρ εγκρίνεται. 171 και 10 είναι ταυτόσιμες. Ποιος είναι υπέρ? Εγκρίνεται. 172 υπέρ. Εγκρίνεται. 173 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 174 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την 174. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Εκατόν εβδομήντα πέντε. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. εφτά υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 178 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 179 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 12 του εισηγητή και 7 ένβη υπέρ, εγκρίνεται. 180 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 182 υπέρ, εγκρίνεται. 183 υπέρ, Εγκρίνεται. 185. ογδόντα Κατά. ηλεκτρονική επαλήθευση για την 185. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. 15 του εισηγητή. Υπέρ. Εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην τελική ψηφοφορία για την πρόταση όπως τροποποιήθηκε. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται τώρα η ψηφοφορία για το σχέδιο όπως τροποποιήθηκε. Πέρας. Εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην ψηφοφορία για το νομοθετικό ψήφισμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Σας παρακαλώ να ψηφίσουμε τώρα για το νομοθετικό ψήφισμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων χρειάζονται τουλάχιστον 23 θετικές ψήφοι και άρχεται τώρα η επίσης ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας. Μάλιστα, εγκρίνατε. Θα ήθελα τώρα να συγχαρώ τον κύριο Νταντάν. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Κύριε Νταντάν, θα θέλετε να μιλήσετε. Στις 8 θα αρχίσει η συνεδρίαση με τον Επίτροπο. Κάνουμε τώρα 5 λεπτό διάλειμμα και επιστρέφουμε ακριβώς στις 8. Σας ευχαριστώ πολύ για την γρήγορη και αποτελεσματική ψηφοφορία.

Αγαπητοί συνάδελφοι, ας περάσουμε τώρα στο δεύτερο τμήμα της συνεδρίασής μας. Θα ήθελα λοιπόν να καλωσορίσω στην Επιτροπή μας τον Επίτροπο Φιλ Χόγκαν, τον δικό μας τον Επίτροπο, Θα θυμάστε ότι το 2013 εγκρίθηκε μια νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δάση και στη συνέχεια είχαμε και τη δική μας έκθεση πρωτοβουλίας από την κυρία Κέστιγκερ και η έκθεση αυτή όπως θα θυμάστε εγκρίθηκε με πολύ μεγάλη πλειοψηφία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στην έκθεση αυτή γίνεται σαφής μνήα για την ανάγκη μιας σφαιρικής προσέγγισης όσον αφορά τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δάση και αναφερθήκαμε επίση και στην ανάγκη για τον κατάλληλο συντονισμό ανάμεσα στα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ολομέλεια, μάλιστα, τότε ο Επίτροπο μα είχε πει ότι θα ερχόταν να μα δει εδώ, στην Επιτροπή μα, προκειμένου να μα μιλήσει λίγο για τη διαδικασία εφαρμογή αυτή τη στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση για τα δάση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ένα πολιτέ σχέδιο εφαρμογή για τα δάση και τη δασική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δημοσιοποιήθηκε το Σεπτέμβριο το κείμενο αυτό. Και όντω, όπω βλέπετε, ο Επίτροπο κράτησε τι υποσχέσει του και όντω έχει έρθει εδώ πέρα να μα μιλήσει για αυτό το σχέδιο εφαρμογή, το πολιτέ σχέδιο εφαρμογή όσον αφορά τη δασική στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ελπίζω, θέλω να ελπίζω, ότι θα αναφερθεί επίσης και στα επιμέρους προγράμματα τα οποία έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο αυτού του πολιετούς σχεδίου εφαρμογή, το αποκαλούμενο Forest Map. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή να αναφερθούμε στο σύνολο του εγγράφου. Δεν πρόκειται τουλάχιστον εγώ να το κάνω σε καμία περίπτωση. Πρόκειται για έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής άλλωστε. Θα δώσω καταρχάς το λόγο λοιπόν στον Επίτροπο και στη συνέχεια στους συντονιστές της Επιτροπής μας και στη συνέχεια σε οποιονδήποτε άλλο ενδεχομένως θέλει να πάρει το λόγο. Κυρίες και κύριοι, το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον αλλά σας παρακαλώ πολύ ας επικεντρωθούμε πραγματικά στο ζήτημα αυτό και εμείς ακουμπήσουμε άλλα ζητήματα. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ για να σας παρουσιάσω το πολίτες εφαρμοστικό ε, πρόγραμμα για την στρατηγική για τα δάση Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ήθελα να αναφερθώ και στους ε, επιτρόπους Ζέσσα και Βέλα που συμμετείχαν πολύ δραστήρια σε όλη αυτή την προσπάθεια. Εμείς Συνεργαστήκαμε με τα κράτη-μέλη και λάβαμε υπόψη και τα όσα μας δήλωσαν οι εμπλεκόμενοι φορείς από το χώρο της δασοκομείας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη χάραξη αυτής της στρατηγικής. Χαιρετίζω τις εργασίες αυτής της Επιτροπής και την ε, γνωμοδότηση πρωτοβουλίας και θα ήθελα να αναγνωρίσω τα όσα έκανε η συγγήτρια κυρία και όπως επίσης και οι σχεδόντες συγγητές. Γνωρίζουμε πως η ευρωπαϊκή κοινωνία ε, πιστεύει στα δάση. Είναι μία από τις βασικότερες χωροταξικές χρήσεις. Είναι το 40% της ε, έκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επεκτείνονται. Τα δάση είναι ένας πολύ σημαντικός οικονομικός κλάδος, έτσι ώστε οι περιοχές της Υπέθρου να είναι ζωντανές, να είναι βιώσιμες. Πάνω από 3 εκατομμύρια θέσεις εργασίας προσφέρουν και είναι ένα ουσιαστικό ε, στοιχείο για τη διατήρηση της χλωρίδας πανίδας και οικοσυστήματος στην Ευρώπη. Τα δάση προστατεύουν την βιοποικιλότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προσφέρουν πολλές υπηρεσίες στα σχετικά οικοσυστήματα. Είναι ένας κομβικός κλάδος στη μετάβαση προς μια οικονομία η οποία είναι φιλική προς το περιβάλλον και χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Αυτή τη στιγμή έχουμε περισσότερες ευκαιρίες παρά προκλήσεις. Χρειαζόμαστε όλο και μεγαλύτερες, ε, μεγαλύτερα αποθέματα βιομάσας. Αυτό και λόγω των εξελίξεων στην ε, παγκόσμια οικονομία. Επίσης τα οικοσυστήματα ε, αντιμετωπίζουν κινδύνους πλήττονται από ξηρασία, από φωτιά ε, δασικές πυρκαγιές και από νέα παράσιτα που τα καταστρέφουν. Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να αναπτύξουμε τα δάση έτσι ώστε να έχουμε μια ισόρροπη ανάπτυξη που θα, επιτρέψει τα δάση να επιβιώσουν παρόλες τις απειλές που θα συναντούν. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε μέσα τη στρατηγική μας. Συγκεκριμένοι στόχοι να ενισχύσουμε τις ε, ε που κάνουμε για τη μείωση της αποψήλωσης παγκοσμίως, όπως επίσης και για να έχουμε βιώσιμη ε, στρατηγική για τα δάση. Να ακολουθούμε τις σωστές πρακτικές και αρχές και υπενθυμίζω το ψήφισμα του Κοινοβουλίου που μας ζήτησε η εφαρμογή της ε, στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γίνει μέσω ενός συντονισμένου πολιετούς πλησίου με αποτελεσματικό τρόπο, με συνέπεια και με την ελάχιστη δυνατή ε, την ελάχιστη δυνατόν γραφειοκρατία. Όλα αυτά τα στοιχεία θα τα βρείτε στο σχέδιο δράσης και εφαρμογής που παρουσιάζουμε και αυτά είναι ε, σε απόλυτη συνέπεια με την δική μου δέσμευση για απλούστευση και σε άλλους χώρους, με συγκεκριμένες δράσεις. Με τσι, το σχέδιο αυτό θα οδηγήσει εμάς και τον κλάδο στο να πετύχουμε τους στόχους του 2020 και ε, στο, να ανταποκριθούμε στις διάφορες προτεραιότητες που έχουμε χαράξει. Συνέπεια, συνοχή, συντονισμό των διαφορών πολιτικών για τα δάση, και πιο συγκεκριμένα λαμβάνοντας υπόψη τους εμπλεκόμενους φορείς. Ο συντονισμός αυτός είναι όλο και πιο σημαντικός δεδομένων των αποφάσεων που θα πρέπει να ληφθούν ε, στην Σύνοδο ε, τη σχετική και για τα χωροταξικά θέματα τα οποία θα δούμε εν ώψη του πλαισίου για την ενέργεια για το 2030. Επίσης θα πρέπει να έχουμε βιώσιμα βιοκάψιμα και βιομάζα που έχουμε πει ότι θα εντάξουμε στο πακέτο για τι ανανεώσιμε 2016 2016-2017 και για μια προπράσινη οικονομία. Όπω αναφέρεται στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το πολιτέ αυτό σχέδιο αναγνωρίζει την ανάγκη να θέσουμε προτεραιότητε που θα είναι η ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα των ε, δασών. Να στηρίξουμε τι ε, περιοχέ τη υπαίθρου και να ευθυγραμμιστούμε με τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές που μας έχει δώσει ο πρόεδρος κ. Γιούγκερ. Γιατί ξέρετε πως ο κλάδος της νοσοκομείας είναι το 7% περίπου ε, του ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προσφέρει πάρα πολλές θέσεις εργασίες στις υπαίθριες περιοχές όπου οι ευκαιρίες αυτές είναι μάλλον σπάνιες δασική βιομάζα και αυτό σημαίνει πως ο κλάδος έχει περιθώριο να αναπτυχθεί πολύ περισσότερο και να συνεισφέρει και στην ε, ατζέντα για την ανάπτυξη και για την απασχόληση. Το σχέδιό μας προωθεί ε, την χρήση του ξύλου ως βιώσιμο και ανανεώσιμο προϊόν ενέργειας για να έχουμε μια η οικονομία η οποία θα βασίζεται σε πιο ευέλικτες μορφές ενέργειας. Το σχέδιό μας τονίζει επίσης πως πρέπει να υπάρχει συνέπεια μεταξύ των διαφόρων εργαλείων πολιτικής που θα χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή. Τα προγράμματα ανάπτυξης, αγροτικής ανάπτυξης προσφέρουν ευκαιρίες στα κράτη-μέλη, επενδύσεις, προώθηση, εμπόριο, ε, στήριξη των ενώσεων παραγωγών, ε, και πρέπει να σας πω πως στα ε, προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης που έχουν ήδη εγκριθεί και στις προτάσεις στα 31 που δεν έχουν εγκριθεί δώσαμε 7,2 δις για την περίοδο 2014-2020 στα δάση το ετήσιο πρόγραμμα θα εξολογήσει πώς μπορούν αυτά να δώσουν προσθέμενη αξία, πώς μπορούν να εφαρμοστούν πιο αποτελεσματικά. Εμείς αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να δημιουργήσουμε και ένα χρηματοπιστωτικό εργαλείο που θα επιτρέπει τα κράτη-μέλη να χειριστούν τα δασικά θέματα μέσω και της ΕΤΕ, μέσω και του χρηματοδοτικού μηχανισμού και πιστεύουμε πως αυτό θα είναι ε, πολύ σύντομα στη διάθεσή σας. Έχουμε ένα ακόμα εργαλείο για την εφαρμογή που είναι το 7ο πρόγραμμα δράση για το περιβάλλον. Αναθεωρεί το πλαίσιο για την καλύτερη διαχείριση του περιβάλλοντος. Αυτό με ικανοποιεί ιδιαίτερα γιατί εγώ διαπραγματεύτηκα τη στρατηγική αυτή με το Κοινοβούλιο και ε, με το Συμβούλιο στα πλαίσια της Ιρλανδικής Προεδρίας το 2013. Έχουμε το Horizon 2020, έχουμε την εταιρική σχέση για την έρευνα. Αυτά θα στηρίξουν οικονομικά τον κλάδο στο μέλλον και κυρίως την βιοοικονομία που θα βασίζεται σε ΣΒΙΤ. Το πρόγραμμα το πολιετές για τα δάση ασχολείται και με κάποια παγκόσμια θέματα. Εμείς είμαστε ε, στις επάλξεις προσπαθώντας ε, καταρχήν ε, να δούμε πώς μπορούμε να επιβάλλουμε το σχέδιο δράσης για τη διαχείριση των δασών, πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε την αποψήλωση, ε, την αποδάσωση και πρέπει να σας πω πως επόμενα βήματα είναι η διατύπωση ενός ετήσιου προγράμματος και μια ενδιάμεση αναθεώρηση εν ώψη του 2020. Ξέρετε πως τα δάση είναι πολύ διαφορετικά σε διάφορα κομμάτια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε έχουμε την αρχή έτσι ε, επικουρικότητας, της καλύτερης νομοθεσίας και της αναλογικότητας που θα αποτελέσουν τον πυρήνα του προγράμματος. Για την εφαρμογή της νέας στρατηγικής πρέπει να σας πω πως η συμφορά σας είναι ιδιαίτερα καλοδεχόμενη. Θα σας ενημερώνουμε για την πρόοδο, για τις συγκεκριμένε δράσεις και θα πω και δύο λόγια στο τέλος αφού ακούσω τα όσα εσείς θα σχολιάσετε. Dziękujemy panie komisarzu. Tak jak zapowiedziałem, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Όπως ανακοίνωσα και νωρίτερα, θα λάβουν το λόγο τώρα οι εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων και για το ΕΛΚ έχει το λόγο πρώτο η κυρία Κώστινιαρ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μας δώσατε να σας ακούσουμε σήμερα. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, η δασική στρατηγική. Και εμείς εδώ στην Επιτροπή έχουμε επεξεργαστεί πάρα πολύ διεξοδικά το θέμα, έτσι ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει μια σαφή θέση για την δασική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως αναφέρατε ήδη, τα δάση είναι πολύτιμα, πολύτιμα και για την οικονομική ανάπτυξη και για την ε, ενεργειακή ε, ανάπτυξη και είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε το δυναμικό που μας δίνουν τα δάση ε, σε όλη του την έκταση. Χαίρομαι πάρα πολύ που δίνεται ιδιαίτερη αξία στην ε, δασική στρατηγική και την θεωρείται κινητήριο δύναμη έτσι ώστε να αυξηθεί η παραγωγικότητα και επίσης που μιλήσετε για τη μείωση της γραφειοκρατίας. Επίσης ε, μην ξεχνάμε την ε, οικονομική, την οικολογική κυρίως σημασία των δασών για την Ευρώπη. Θα ήθελα να σταθώ σε ένα σημείο το οποίο έχουμε συζητήσει διεξοδικά σε αυτήν εδώ την Επιτροπή, δηλαδή την συμπερίληψη των ιδιοκτητών των δασών, ιδιαίτερα ε, των όσων διαχειρίζονται οικονομικά τα δάση. Έχουμε αναφέρει έντονα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει μία αρμόδια επιτροπή και μία αξιολόγηση αυτής. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση και τι σχεδιάζει να κάνει. Βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία όλο ένα και περισσότερο ε, προσπαθεί να ε, αποδυναμώσει την ε, ισχύ των ιδιοκτητών των δασών. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να δούμε και την ε, οικονομική τους αξία, να δούμε και την εμπειρογνωμοσύνη που διαθέτουν οι ιδιοκτήτες των δασών και όσοι τα εκμεταλλεύονται οικονομικά και να συμπεριληφθούν και εκείνοι υπόψη στην δασική στρατηγική. Επίσης, ε, θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής, ε, πόσο έχουν προχωρήσει τα σχέδιά σας έτσι ώστε να μπορέσουμε να συνεργαστούμε μαζί σας ε, όσο το δυνατόν καλύτερα. Θα θέλαμε να μας ενημερώνετε φυσικά. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ντεκάστρο έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που ήρθατε εδώ στην Επιτροπή μας και που μπορούμε να κάνουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Ξέρω ότι είχαμε συζητήσει και το πρόγραμμα Juncker στο παρελθόν. Ξέρουμε ότι η στρατηγική αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική. Η κυρία Κέστιγκερ μας είπε πόσο σημαντική είναι η στρατηγική αυτή. Σίγουρα πάντως ε, θα θέλαμε να μπορούμε να είχαμε και έναν διάλογο μαζί σας προκειμένου να συζητήσουμε τις τόσες δυσκολίες, την κρίση αυτή που πλήττει πραγματικά τον αγροτικό κόσμο στην Ευρώπη. Και πρέπει να πούμε ότι όσον αφορά την ζωοτεχνική νομοθεσία. Είχατε εσείς μια πολύ σημαντική και γρήγορη παρέμβαση, αλλά θα μπορούσαμε να αποδοκιμάσουμε κάποια σημεία της στρατηγικής σας. Για παράδειγμα, όσον αφορά τον κανονισμό για το γάλα και τα φρούτα στα σχολεία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ζητήσει να διατηρηθεί ο κανονισμός αυτό στο θεματολόγιο εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτό που ακούμε τώρα είναι ότι υπάρχουν πολλές χώρες που θέλουν να αλλάξουν την νομική βάση και να αποκλείσουν τελικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την δυνατότητα συναπόφασης που έχει στο συγκεκριμένο αυτό φάκελο. Εμείς προφανώς αποδοκιμάζουμε κάτι τέτοιο και θα θέλαμε να συνεχίζεται ως εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υποστηρίζει στηρίζεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Κύριε Μίλλερ, έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση αυτή. Η εφαρμογή της δασικής στρατηγικής παίζει έναν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για τους ε, ιδιοκτήτες των ε, δασών της Ευρώπης και η τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, είναι κάτι που θα συνεισφέρει πολύ σημαντικά στις ε, περαιτέρω εξελίξεις. Την περασμένη εβδομάδα η παρευρέθησα στην απονομή του βραβείου για τα δάση και εκεί συμμετείχαν πάρα πολλοί ιδιοκτήτες μικρών δασικών εκτάσεων και με ενημέρωσαν σχετικά με τα σχέδια εκμετάλλευσης των δασών, τα οποία εσείς έχετε απορρίψει. Θα ήθελα λοιπόν ε, να πω πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να δείξει θάρρος και εμπιστοσύνη στους ε, ιδιωτικούς φορείς που διαχειρίζονται και εκμεταλλεύονται τα δάση, διότι εκείνοι έχουν το ε, καλό των δασών ως κύριο μέλημά τους. Επίσης, ε, αναφερθήκατε στην λιγότερη γραφειοκρατία. Αυτό είναι αναγκαίο σε όλους ε, τους τομείς και σε όλα τα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο παρατηρώ πως ε, υπάρχουν προβλήματα στη γωνία ιδιαίτερα όταν ε, μας αναφέρατε ότι στα πλαίσια του ορίζοντα 2020 υπάρχουν ορισμένα κονδύλια. Δεν μπορώ να δω όμως ε, από αυτά τα δισεκατομμύρια ευρώ που βρίσκονται στο πρόγραμμα ορίζοντας 2020 κάποια ε, προγράμματα που να αφορούν τη διαχείριση των ε, δασών και φοβάμαι πολύ ότι θα ζημιωθούν στο τέλος και οι τοπικές κοινωνίες και οι ιδιοκτήτες μικρών δασικών εκτάσεων που διαχειρίζονται οικονομικά τις εκτάσεις αυτές. Μιλάμε για μικρές ε, κοινότητες ε, ανθρώπων οι οποίοι ζουν από τα δάση και όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει κάποιο ε, σχέδιο που να τους συμπεριλαμβάνει αλλά αντίθετα παρεμβαίνει στην ιδιοκτησία τους τότε αυτό είναι ζημιογόνο. Ε, κύριος έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Η σημασία της ε, δασοπονίας στην Ιρλανδία ήρθε στο προσκήνιο περίπου όταν ανέβηκε στην εξουσία και η τωρινή μας κυβέρνηση. Έγινε μια συζήτηση για το αν όλα τα δάση θα έπρεπε να ξεπουληθούν για να ξεπληρώσουμε τα χρέη που επομιστήκαμε. Έγινε λοιπόν μια συζήτηση για το θέμα αυτό και η συζήτηση αυτή οδήγησε σε ε, αύξηση του ενδιαφέροντος από εκείνους που ήδη βρίσκονταν στον ε, χώρο αυτό της δασικής εκμετάλλευσης. Δυστυχώς όμως με αρνητικές επιθανές συνέπειες σε καταστροφή του περιβάλλοντος κτλ. Στο τέλος καταφέραμε να ε, κάνουμε σαφές ε, το πόσο επικίνδυνη ήταν αυτή η πρόταση και δεν πουλήθηκαν τα δάση. Θα ήταν τρέλα να πουληθούν τα δάση στην Ιρλανδία. Έχω λάβει πολλές ε, πληροφορίες από εταιρείε που διαστηριοποιούνται στον ε, τομέα της δασοπονίας και μια κρατική εταιρεία μάλιστα από ό,τι γνωρίζω διαχειρίζεται την ε, πλειοψηφία των δασών. Γι' αυτό κύριε Επίτροπε ήθελα να σας ρωτήσω θα, θα μπορέσετε εσείς να μας βοηθήσετε. Έχουμε πολλές κατηγορίες για περιπτώσεις απάτη και βλέπω πως ε, προσπαθείτε μεν να προφυλάξετε τα δάση στην Ευρώπη, αλλά δεν κάνατε τίποτα για τα δάση της Ιρλανδίας. Τα δάση το τελευταίο που χρειάζονται είναι ε, διαχειριστικούς φορείς που τα εκμεταλλεύονται και που εξαπατούν. Δυστυχώς αυτός ο ή μη οργανισμός που τα διαχειρίζεται δεν ε, δέχεται να συνεργαστεί. Τώρα όμως έχουμε έναν επίτροπο αρμόδιο για αυτό το θέμα στην, από την Ιρλανδία, από τη χώρα μου. Γι' αυτό λοιπόν κύριε επίτροπε, εάν εγώ έρθω σε εσά με αυτές τις πληροφορίες που έχω στη διάθεσή μου, θα μπορέσετε να κάνετε κάτι γι' αυτό. Έχουμε πληροφορίες για απάτη ύψους 80 έως 90 εκατομμυρίων ευρώ από αυτούς τους ε, ημικρατικούς οργανισμούς. Θα ήθελα λοιπόν να μάθουμε εάν, αυτό, ε, αν αυτές οι κατηγορίες αληθεύουν και αν αληθεύουν θα πρέπει να δράσουμε. Δυστυχώς ο τομέας της δασοπονίας ε, δεν επωφελείται καθόλου, διότι η πλειονότητα των ε, ε, φορέων που διαχειρίζονται και εκμεταλλεύονται οικονομικά τα δάση αρνούνται να συνεργαστούν μαζί μας για την προστασία τους. Εσείς θα μπορέσετε να κάνετε κάτι γι' αυτό. Ο κύριος Χόισλινγκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, πολύ ωραία που ήρθατε. Όμως αναρωτιέμαι εάν πρέπει να περιοριστούμε μόνο στην ε, δασοπονία. Είναι τόσο πολλά τα θέματα που θέλουμε να συζητήσουμε μαζί σας. Γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο να περιοριστώ σε αυτό. Θα ήθελα να σταθώ σε μία συνέντευξη που δώσατε την περασμένη εβδομάδα. Μας αναφέρατε τους ε, γαλακτοπαραγωγούς και αρνηθήκατε το γεγονός ότι υπάρχει κρίση παρά το, τα στοιχεία που αποδεικνύουν το αντίθετο. Η κρίση στην αγορά των, της επαγωγής γάλακτος ε, απειλεί το βιός πάρα πολλών εργαζόμενων στον τομέα αυτό. Και πραγματικά αναρωτιέμαι εάν έχετε αναγνωρίσει ότι υπάρχει κρίση, διότι μου φαίνεται το αντίθετο. Και βλέπω ότι Υπάρχει σύγκρουση ενδιαφέροντος ανάμεσα στους χρήστες και οικονομικούς αφορείς που διαχειρίζονται τη βιομάζα και ε, σε όσους θέλουν να προστατεύσουν το περιβάλλον. Το γεγονός είναι ότι υπάρχουν προβλήματα σε όλους ε, τους ε, τομείς της γεωργίας, υπάρχουν προβλήματα στην δασοπονία βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές ε, υπερβολικά ε, υψηλές εξαγωγές στρογγυλής ξυλίας προς την Κίνα. Μάλιστα έχουν πενταπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια. Θα μπορούσατε εσείς ε, να μας πείτε εάν πραγματικά υπάρχει κάποιο πρόβλημα σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων ή όχι. Επίσης, θεωρείτε πως η νομοθεσία για το δίκτυο Natura 2000 χρειάζεται αναθεώρηση χρειάζεται διόρθωση. Εγώ θεωρώ πως ε, η νομοθεσία για το δίκτυο Natura έχει προσφέρει πολλά για την προστασία των δασών. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Άγνιου έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Νομίζω ότι πάντα φαίνεται να υπάρχει ένα είδο ε, συνωμοσία, ε, κάποιο σενάριο το οποίο υποθάλπει κάθε φορά που έρχεται ο Επίτροπος εδώ πέρα να μας δει και πάντα εκφράζονται απόψε αυτέ από την ε, Ιρλανδική αριστερά, από τον κύριο Φάναγκαν. Πάντω ο συνήθως και εγώ θα συμβάλλω κατά τον ίδιο τρόπο. Αν κατάλαβα καλά, σύμφωνα με τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν θα έπρεπε κανονικά να γίνεται συνεδρίαση της Επιτροπής μας εδώ πέρα στο Στρασβούρο κάτι διάρκεια της Ολομέλειας. Ενδεχομένως να έχουν γίνει κάποιες αλλαγές και να μην τις γνωρίζω. Το πιο σημαντικό πάντως είναι ότι ανέκαθεν η δασοπονία δεν αποτελούσε αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Γεωργία σίγουρα ναι, αλλά από όσο γνωρίζω μου λένε ότι η δεσοπονία δεν εμπίπτει σε αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όταν μας λέει λοιπόν ο Επίτροπος ότι θέλει να μειώσει τη γραφειοκρατία, όλοι προφανώς είμαστε υπέρ κάτι τέτοιου, δεν θα έπρεπε να υπάρχει καμία γραφειοκρατία πουθενά, αλλά θα μεταφέρω εγώ ουσιαστικά την πληροφορία αυτή στου υπεύθυνου για τη δασοπονία στη δική μου τη χώρα, οι οποίοι θα νομίζουν τελικά ότι ο επίτροπο είναι αρμόδιο όντω για τη δασοπονία. Αναφερθήκατε επίση στην κλιματική αλλαγή, το νέο όρο που χρησιμοποιούμε για την υπερθέρμανση του πλανήτη που τελικά δεν έλαβε χώρα. Κόβουμε όλα αυτά τα δέντρα, δημιουργούμε βιομάζα και αυτό λειτουργεί θετικά, όπω μα είπατε. Εγώ από εμπορική πλευρά ασχολήθηκα με το τομέα αυτό και έχασα πάρα πολλά χρήματα, γιατί κοστίζει τελικά πολύ περισσότερο το να κόψει κανεί τα δέντρα αυτά, να τα μεταφέρει στι καταστάσεις εκείνες που θα μετατρέψουν σε βιομάζα και ουσιαστικά από οικονομικής πλευράς μπορώ να πω ότι ζημιώθηκα. Και νομίζω ότι ε, θα έπρεπε να χαιρόμαστε όλοι που αυξάνονται οι εκπομπές εξωτερικού του άνθρακα, γιατί αυτό σημαίνει ότι θα αυξηθούν, θα μεγαλώσουν πολύ πιο γρήγορα τα δέντρα. Επομένω, ουσιαστικά δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας έτσι δεν είναι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, Νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε τώρα το λόγο στον Επίτροπο για να απαντήσει όλες αυτές τις ερωτήσεις. 26 είναι συνολικά οι ομιλητές που θέλουν να πάρουν το λόγο. Επομένως μιλήσει παρακαλώ πολύ για 1,5 το πολύ 2 λεπτά προκειμένου να δώσουμε και τη δυνατότητα στον Επίτροπο να απαντήσει σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Μην υπερβείτε το χώρο της ομιλίας, μην μιλάτε πάνω από δύο λεπτά. Θα ακούσουμε λοιπόν τις ερωτήσεις και θα μπορέσει στη συνέχεια να απαντήσει ή να σχολιάσει ο Επίτροπος. Η κυρία Χέρνης Γκαρσία έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο που ήρθε να μας επισκεφθεί απόψε και βεβαίως τα όσα είπε η κυρία Κόστιγκερ τα προσπογράφω και εγώ. Είναι πολύ σημαντικό και χρειαζόμαστε μια σφαιρική προσέγγιση. Αυτό είναι απαραίτητο, αλλά πρέπει να είναι ευρωπαϊκή αυτή η στρατηγική, γιατί τελικά είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών και κυρίως αν ε, περάσουμε από το δεύτερο πυλώνα της ε, ε, Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για τη χρηματοδότηση. Ξέρετε πως για την αγροτική ανάπτυξη στη χώρα μου για παράδειγμα αρμόδιες είναι οι περιφέρειες και έχουν την επιλογή. Άρα λοιπόν θα πρέπει αυτό να το λάβουμε υπόψη και αν θέλουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό τότε μιλάμε και για άλλου είδους χρηματοδότηση, άλλου ύψους. Τι σημαίνει αγροτική ανάπτυξη τι σημαίνει αυτή η στρατηγική που έχουμε, γιατί για να τα συνδυάσουμε με τον τρέχοντα προπολογισμό σα έχουμε δυσκολίε Στην επιστολή του ε, κυρίου Γιούγκερ τη προηγούμενη εβδομάδας, ε, που μιλάμε για απλούστευση, για τις δημοσιονομικές ε, προοπτικές, μιλά για κάποια για επαναπροορισμό, επαναπροορισμό της κοινή αργετικής πολιτικής. Τι σημαίνει αυτό. Θα μιλήσουμε για οικονομική μεταρρύθμιση το 2016 της ΚΑΠ ή θα περιμένουμε το 2018 για να το κάνουμε. Είναι πολύ σημαντικό το στοιχείο αυτό και όλοι οι παραγωγοί ε, είτε είναι κτηνοτροφικά είτε γεωργικά είτε δασικά προϊόντα ανησυχούν ιδιαίτερα στη χώρα μου για το θέμα αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Μπράνον παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είμαστε υπέρ του σχεδίου αυτού εφαρμογή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βλέπουμε ότι αντέδρασε πολύ γρήγορα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τα όσα συζητήσαμε εδώ στο Κοινοβούλιο. Και νομίζω είναι θετικό το ότι βλέπουμε ότι συνειδητοποιεί τελικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη σημασία που έχουν τα δάση και η ξυλία στην καταπολέμηση τη κλιματική αλλαγή. Πρόσφατα είχα πάει στη Νότιο Γαλλία μαζί με έναν συνάδελφό μου και είδαμε πραγματικά τον ε, ρόλο που μπορεί να παίξουν τα δάση και στην απορρόφηση διοξιδίων, ε, εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και στην διατήρηση του εδάφους και στην καταπολέμηση της διάβρωσής του. Τρεις σύντομες παρατηρήσεις όσον αφορά την χρήση της γης, το LULUCF, χρήση γης, αλλαγή στη χρήση γης, δαξικομικές δραστηριότητες. Πώς πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να ενταχθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια. Νομίζω ότι θα πρέπει να προσδιορίσουμε σωστά τα πράγματα, το οποίο θα είναι θετικό. Αν όμως κάνουμε λάθη στις μετρήσεις μας, τα πράγματα θα είναι προβληματικά. Πώς μπορεί λοιπόν η χρήση γης και η αλλαγή της χρήσης γης να σωματωθεί στο ζήτημα του κλίματος και της ενέργειας. Δεύτερη παρατήρηση, ζήτημα το οποίο έθιξαν και οι συνάδελφοι πριν από λίγο. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης βλέπουμε ότι έρχονται πάρα πολλές μεγάλες ποσότητες βιομάζας από τη Βόρεια Αμερική. Ποια είναι η δική σας η προσωπική άποψη. Νομίζω ότι πραγματικά είναι τεράστια η απόσταση αυτή που πρέπει να διανυθεί τελικά για να κάψουμε στην Αγγλία πριν ήδη που έρχεται από την, ΗΠΑ. τις Πιστεύετε ότι είναι βιώσιμο να κάνουμε τελικά κάτι τέτοιο. Και τρίτον, είναι πολύ σημαντικό από κοινού να συντοπίσουμε ότι υπάρχουν κάποια υγειονομικά ωφέλη τα οποία μπορούν να προκύψουν από τα δάση. Λυπάμαι που θα πρέπει να αποχωρήσω γιατί πρέπει να μιλήσω στην Ολομέλη και ενδεχομένω να μην ακούσω την απάντησή σας. Πρέπει να πάω στην Ολομέλη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ έχω ερωτήσει για εσά, κύριε Επίτροπε. Θα μπορούσαμε να μιλάμε όλο το βράδυ για τα δάση, γιατί είναι κάτι τόσο σημαντικό, το οποίο αξίζει τόσο ε, μακροχρονία συζήτηση. Καταρχά, να ρωτήσω. Είστε υπέρ τη ε, χρήση, της ε, έντονης εκμετάλλευσης ε, της ε, ξυλίας στην Ευρώπη. Έπειτα, Αναφέρετε στην ε, παρουσίασή σας ότι πρέπει να υπάρχουν κριτήρια αηφορίας. Υπάρχουν κάποια δεσμευτικά κριτήρια αηφορίας για όλη την Ευρώπη. Αυτό θα ήθελα να το μάθω. Επίσης, θα ήθελα να μάθω εάν δάση τα οποία ανήκουν στο κράτος, ε, στο δημόσιο δηλαδή, θα ε, εκμεταλλεύονται οικονομικά από εδώ και στο εξή ε, με τρόπο υποδειγματικό. Εσείς ως Επίτροπος ε, Γεωργίας θα μπορούσατε να επηρεάσετε, να την ε, αηφόρο διαχείριση των ε, δασών που ανήκουν στο δημόσιο. Επίσης υπάρχουν ζημιές που παθαίνουν τα δάση και αυτές προκαλούνται όχι από πυρκαγιές αλλά από τα άγρια ζώα. Θα ήθελα να μάθω την άποψή σας σχετικά με αυτό. Επίσης αναφέρατε στην παρουσίασή σας πως υπάρχει τεράστιο δυναμικό στα δάση. Τα δάση όμως δεν είναι ατελείωτα. Υπάρχουν ε, κατά τη γνώμη σας όρια στην χρήση, στην οικονομική εκμετάλλευση των δασών. Πρέπει να υπάρχουν όρια. Και τέλος, ε, για το μόνιμο συμβούλιο για τα δάση. Είπατε πως ε, θα συμπεριλαμβάνονται εκπρόσωποι από όλους τους φορείς και θα αυξάνονται τα μέλη αυτού του Συμβουλίου. Εγώ θα ήθελα να μην αυξάνονται εσάι e τα μέλη, αλλά να αυξάνονται ε, ποιοτικά, όχι ποσοτικά. Είναι στο χέρι σας, ε, κύριε Επίτροπε, να σώσετε τα δάση και έχετε τεράστια ευθύνη γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Νέκοφ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, μα ζητήσατε να είμαστε σαφείς και θα το προσπαθήσω. Πριν όμως θα ήθελα να σας συγχαρώ για το πολιετές πρόγραμμα εφαρμογής της δασικής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαίρομαι που είπατε ότι τα δάση δεν είναι μόνο ξυλία, αλλά είναι και σημαντικά για τη βιοπικιλότητα. Επισκεφθήκατε τη χώρα μου, τη Βουλγαρία και είδατε με τα μάτια σας ότι τα βότανα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Εμείς συλλέγουμε βότανα τα οποία φυτρώνουν στα δάση, μανιτάρια, ε, διάφορα είδη φυτών και νομίζω ότι αυτή η συλλογή η συγκομιδή βοτάνων θα μπορούσε να είναι μια σημαντική πηγή απασχόλησης για τους κατοίκους ε, των ε, περιοχών αυτών. Βότανα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ε, παρασκευή καλλιντικών, για παράδειγμα. Έχω λοιπόν την εξή ερώτηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν νομίζετε πως χρειάζεται μια στρατηγική σχετικά με τα βότανα. Ίσως η συλλογή βοτάνων θα μπορούσε να συνεισφέρει οικονομικά στην ανάπτυξη και είναι κάτι που είναι επίσης ε, πολύ σημαντικό για τη βιοπικιλότητα. Ο τρόπος με τον οποίο συλλέγονται τα βότανα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικό για την διατήρηση των φυτών αυτών. Διαφορετικά τα αποτελέσματα θα είναι καταστροφικά. Όπως σας είπα, η πρακτική αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική, ιδιαίτερα μάλιστα στα πλαίσια όσων αναφέρεται για ε, την βιοοικονομία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα κύριε Πίτροπε να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που βλέπουμε ότι τροποποιήθηκε ένα λόγο ημερήσια διάταξη τη ε, συνεδρίασή μα και όπω και στην αδερφή μου, θεωρώ και εγώ ότι η στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τα δάση είναι πολύ σημαντική στα πλαίσια τη ανάπτυξη τη υπαίθρου. Έχω μόνο ένα λεπτό στη διάθεσή μου. Μου φαίνεται λοιπόν περίεργο αυτή τη στιγμή να μιλάμε για μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα σχέδια τη στιγμή που διανύουμε μια πραγματική γεωργική κρίση παντού στην Ευρώπη και τη στιγμή που οι αγρότες μας διανύουν, αντιμετωπίζουν πάρα πολλές αντικσότητες. Και ξέρετε ότι έχουμε αντιμετωπίσει πάρα πολλά προβλήματα όσον αφορά την τιμή του βόλου ή του χείριου κρέατος. Δεν μπορούμε να ξεχνάμε λοιπόν την καθημερινότητα, τις καθημερινές δυσκολίες των γεωργών μας. Δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν υπάρχει κρίση. Όλα αυτά τα βλέπουμε σε καθημερινή βάση, ερχόμενοι σε επαφή με τους γεωργού μας και τους κοινοτρόφους. Νομίζω ότι ο εκπρόσωπος των νέων γεωργών στη Γαλλία σας έχει καλέσει να πάτε να τους δείτε, πρέπει να αντιποκριθείτε στην ε, πρόσκληση αυτή, διότι θα δείτε ότι στην πράξη τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά από ό,τι φαίνονται, από ό,τι συζητάμε εδώ πέρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα πλαίσια τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Όσον αφορά τώρα τα δάση, σε σχέση με αυτά που είπαν οι συνάδελφοι, θα ήθελα και εγώ να θέσω κάποιες, κάποια ερωτήματα. Ποια είναι η δική σας ε, η θέση και εδώ συμφωνώ με τον κύριο Μπράνεν όσον αφορά δηλαδή τη συμβολή των δασών όσον αφορά την κλιματική ε, αλλαγή και την ενέργεια. Και ποια είναι η θέση την οποία εσείς δίνετε όσον αφορά την όλη βιομηχανία των δασών σε σχέση με την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Σελιμόβιτς, κύριε, Σελιμο... Σελιμόβιτς. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κύριε Επίτροπε που ήρθατε και μας προσφέρατε την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί σας. Έχω μια ερώτηση για κάποια περιβαλλοντολογικά στοιχεία που σχετίζονται με τη γεωργία και πιο συγκεκριμένα με τη δασοπονία. Γνωρίζουμε όλοι πως η συνάντηση στο Παρίσι πλησιάζει. Όλοι αναγνωρίζουμε τη σημασία αυτής της συνόδου και όλοι γνωρίζουμε ποια είναι η σημασία της ε, δασοκομείας στη Γεωργία ε, και ποιες είναι οι επιπτώσεις για το κλίμα. Ποιο θεωρείτε εσείς πως είναι τα βασικά εμπόδια και προσκόμματα για μια συμφωνία στο Παρίσι, τουλάχιστον για τα θέματα δασοκομείας και γεωργίας. Να είμαι πιο ανοιχτός. Τι θα θέλατε να δείτε εσείς να εντάσσετε σε μια συμφωνία στο Παρίσι και τι πιστεύετε πως δεν θα μπει στο τραπέζι και σας ευχαριστώ και πάλι που ήρθατε στη συνεδρίασή μας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μποτσόφσκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην Πολωνία τα δάση ανοίγουν στο κράτος και η κοινή γνώμη συμφωνεί απόλυτα με αυτή την ε, κρατική ιδιοκτησία που αποτέλεσε και σημείο τριβής στην προεκλογική περίοδο. Η μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού πιστεύει πως τα δάση θα πρέπει να ανήκουν στο κράτος, στο δημόσιο και να είναι προσβάσιμα από όλους μας. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι κατανοητό. Τα δάση απορροφούν πάρα πολλές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και αυτό κανείς δεν το σκέφτεται παρόλο που αντιμετωπίζουμε την υπερθέρμανση του πλανήτη, την αλλαγή του κλίματος και εμείς προσπαθούμε συνέχεια να κάνουμε χρήση της βιομάζας το οποίο ουσιαστικά μειώνει τις εκτάσεις ε, των δασών ε, και δεν λαμβάνει υπόψη τη σημασία των δασών στην απορρόφηση του δεξιξίδου του άνθρακα. Δεν έχουμε τέτοιου είδους λογική πολιτική και γι' αυτό αμφισβητούμε ε, τις πραγματικές, ε, τους πραγματικούς στόχους όλων αυτών των ε, δράσεων που λένε πως θέλουν να προστατεύσουν τα, το περιβάλλον αλλά ουσιαστικά έχουν κάποιες ε, και καλυμμένες προτεραιότητες. Ο ρόλος των δασών είναι ένα στοιχείο που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη γιατί προστατεύουν το περιβάλλον μας και δυστυχώς αυτό δεν έχει αποτελήσει τον πυρήνα της στρατηγικής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ ο πρόεδρος. Έγινε και μία ακρόαση στην Επιτροπή μας για το θέμα αυτό με πολύ πλούσια στοιχεία που προσφέρθηκαν και κατατέθηκαν από τους συμμετέχοντες. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να τονίσουμε τη σημασία των δασών ως αντίβαρα των περιβαλλοντολογικών μας προβλημάτων και της αλλαγής του κλίματος. Πιστεύω πως αυτό θα ήταν πολύ χρήσιμο και θα έπρεπε να εστιάσουμε σε αυτό. Ίσως δεν αναγνωρίζουμε όλοι ποιο είναι το μέγεθος του προβλήματος το οποίο αναφέρθηκε ο συνάδελφος κ. Βοητσόφσκι. Δηλαδή τα δάση ως καταπολέμηση των προβλημάτων με το κλίμα. Κυρία Αγγιλέρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, εκπλήσωμαι κάπως. Η συζήτηση είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, αναμφισβήτητα. Όμως για τη στρατηγική, τη δασική στρατηγική νομίζω ότι έχουμε κάνει τις δηλώσεις μας, είχαμε τις ανακοινώσεις δικές σας, είχαμε την έκφραση της ε, ε, Ολομέλειας, και νομίζω με τη χρηματοδότηση που βρίσκεται σε κρεμότητα και με τις εγκρίσεις ε, των προγραμμάτων ε, ε, αγροτικής ανάπτυξης που θα στηρίξουν τη χρηματοδότηση νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε φτάσει σε σημείο που να μπορούμε να αξιολογήσουμε το τι γίνεται και όπως λένε οι γεωργοί στη χώρα μας με τα όσα ε, με τα όσα αντιμετωπίζει ο κόσμος ο αγροτικός το να συζητάμε μόνο τα δάση είναι σταγόνα στον ωκεανό όχι ότι δεν είναι σημαντικό αλλά υπάρχουν και άλλα που βασανίζουν τον κλάδο και όπως είπαν αρκετοί συνάδελφοι αυτά τα γνωρίζετε και πάντα είναι μεγάλη χαρά να σας βλέπουμε και οποιοδήποτε θέμα και να συζητάμε αυτό ισχύει αλλά θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία και να σας ρωτήσουμε και για άλλα θέματα και να επιμείνω. Το είπε και η συνάδελφος, η κυρία Ζνάν, υπάρχει κάποια σύγχυση με την επιστολή Γιούνκερ και θα ήθελα να μου πείτε αν θα γίνει αναθεώρηση της ΚΑΠ το 2016 ή το 2018. Πείτε μου, το 16 ή το 18. Γιατί η επιστολή Γιούνκερ και τα λόγια που στη συνόδευσαν δημιουργούν αμφιβολίες. Καλό θα ήταν μια που είστε εδώ μια που έχετε την ευκαιρία να μας ε, ξεκαθαρίζετε το θέμα αυτό, να το κάνετε. Και επίσης, ο νέος κανονισμός ε, για την διανομή γάλακτος και, ε, και φρούτων στα σχολεία. Επίσης πολύ σημαντικό θέμα. Επίσης, ποσόστοση για το ελαιόλαδο, για το ελαιόλαδο. αυξήθηκε η ποσόστοση στην την Ισία πάνω από 3.000 τόνους δίνουμε επιπλέον. Μα εμείς είμαστε παραγωγός χώρο στην Ισπανία και νομίζω ότι καλό θα ήταν να εξηγήσουμε γιατί αυξάνεται η ποσόστοση αυτή για τη χώρα εκείνη και γιατί θα αλλάξουν τα, εξ, τα εισαγωγικά πιστοποιητικά έτσι ώστε να του επιτρέπουν όλο το χρόνο να μας στέλνουν ελαιόλαδο. Υπάρχουν πολλά στοιχεία κύριε Επίτροπε που θα θέλαμε να συζητήσουμε. Θα πρέπει να γίνει μια πιο συνολική συζήτηση. Αλλά τουλάχιστον τι ερωτήσει που σα υπέβαλα σας παρακαλώ να τι απαντήσετε. Κύριε Πατήρ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε. Υπήρξαν πολλές δασικές πυρκαγιές στη χώρα μου. Πολλές πυρκαγιές ε, όπου έκαψαν και δασικές εκτάσεις και αμπέλια. Κόστησαν ε, εκατομμύρια ευρώ σε ζημιές. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από τον Επίτροπο Χόγκαν να μας βοηθήσει να λάβουμε βοήθεια έτσι ώστε να ανανεώσουμε τους αμπελώνες μας το συντομότερο στην Κροατία. Πάνω από το 47% της επικράτειας της Κροατίας αποτελείται από δάση και τα δάση παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για εμάς λοιπόν και για την προστασία του κλίματος. Και εν ώψη του επερχόμενου συνέδριου για το κλίμα, θα ήθελα να ρωτήσω εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει κάποια συγκεκριμένη οικονομική αξιολόγηση της συνεισφοράς των δασών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Οικονομία. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπόγκοβιτς έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλησπέρα σας κύριε Επίτροπε. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω ότι λαμβάνει χώρα για μία ακόμη φορά αυτή η συζήτηση για τα δάση. Η κυρία Κέστιγκερ έχει προτιμάσει μια πάρα πολύ καλή έκθεση και γνωρίζουμε νομίζω όλοι τον σημαντικότατο ρόλο που διδραματίζουν τα δάση. Προέρχομαι από μια χώρα που ένα 60% της επικράτειάς της καλύπτεται από δάση. Και μάλιστα η μάζα της ξυλίας στη χώρα μου αντιστοιχεί σε τεράστιες ποσότητες. Επομένως για τη δική μου τη χώρα ο κλάδος αυτός είναι σημαντικότατος. Επίσης ε, η ποσότητα της ξυλίας που επεξεργαζόμαστε όπως σας είπα είναι πάρα πολύ σημαντική. Και όντω έχουμε συζητήσει σε εθνικό επίπεδο πάρα πολύ τον ρόλο που μπορεί να δραματίσει η δασοπονία. Και σε μια χώρα σαν τη δικιά μου ο ρόλο αυτό μπορεί να είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω περισσότερο ποια μπορεί να είναι η διασύνδεση ανάμεσα στα δάση και την άπτυξη πέθρου. Γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι θα πρέπει να απαντηθεί το ζήτημα αυτό, να διερευνήσουμε περισσότερο τη σχέση αυτή και Κάτι που είναι εξίσου πολύ σημαντικό είναι αυτό το οποίο ονομάζουμε κυκλική οικονομία. Δηλαδή, η ξυλία βλέπουμε ότι δραματίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε όλους τους τομείς της οικονομίας, στον κατασκευαστικό τομέα, στον μεταποιητικό τομέα, στον τομέα της παραγωγής βιοεθανόλης, που μένω στον χημικό επίσης τομέα. Κύριε Πίτροπε, λοιπόν, θα θέλω να κάνω δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις. Πρώτον, Τι προβλέπετε για το μέλλον όσον αφορά την χρηματοδότηση της έρευνας στον τομέα των νέων τεχνολογιών και η χρηματοδότηση αυτή, τα κονδύλια αυτά θα προκύψουν ενδεχομένω και από το Ταμείο Ιούνκερ. Καλησπέρα σας. Εγώ με τη σειρά μου δεν θα σας μιλήσω για δάση, γιατί νομίζω ότι διανύουμε μια πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση σε πάρα πολλές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάρα πολλοί συνάδελφοι αναφέρθηκαν στην κρίση που αντιμετωπίζουν πάρα πολλοί γεωργοί σε πάρα πολλούς γεωργικούς τομείς στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Σαββατοκύριακο αυτό στη Γαλλία ζήσαμε μια πολύ δύσκολη στιγμή. χρειάστηκε να αποτίσουμε για μία ακόμη φορά φόρο τιμή στη Γαλλία στα 600 αυτά άτομα τα οποία αυτοκτόνησαν και αναφέρομαι σε γεωργούς, αγρότες οι οποίοι βρισκόντουσαν σε απόλυτη απόγνωση. Καλείστε λοιπόν εσείς σήμερα να λάβετε μέτρα υπέρ των Ευρωπαίων γεωργών. Μέτρα τα οποία τα ζητάμε εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες κύριε Επίτροπε. Περιμένουμε πλέον από εσά συγκεκριμένες απαντήσεις για να αντιμετωπιστεί η δραματική αυτή κατάσταση που ζούμε. Ačiū pirmininkė, komisarė, už galimybę susitikti. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, είμαι ευγνώμων για το ότι μπορώ να σας κάνω ερωτήσεις σήμερα και έχω κάποιες από αυτές. Όταν η Λιθουανία έγινε ανεξάρτητη το 1990, τα δάση επέστρεψαν στους αρχικούς τους ιδιοκτήτες και στη σήμερα πάνω από το 50% των δασών ανήκουν σε ιδιωτικά χέρια. Το υπόλοιπο ποσοστό ανήκει στο κράτος. όμως δεν υπάρχει αρκετή εμπειρία στην οικονομική διαχείριση των δασών. Εσείς τι άποψη έχετε για την οικονομική συνεργασία στην δασοπονία και ποιες είναι οι μέθοδοι που θα έπρεπε να ε, χρησιμοποιήσουμε. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε βέλτιστες πρακτικές από άλλα κράτη-μέλη ή να στηριχτούμε στην ε, υποστήριξη. Έπειτα, έχω μια άλλη ερώτηση σχετικά με τον γαλακτοπαραγωγικό τομέα. Είναι κρίσιμη η κατάσταση. Έχω συναντηθεί με πολλούς ε, γαλακτοπαραγωγούς και όλοι με ρωτούν το ίδιο πράγμα. Τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για εμάς και τι ε, τι θα απογίνουμε, πώς θα είναι η ζωή μας αύριο με τις ε, αλλαγές που έχουν επέλθει, πόσο μπορούμε να σταματήσουμε την συνεχιζόμενη πτώση της τιμής του γάλακτος. Μπορείτε να μας πείτε κάτι γι' αυτό. Η κυρία Μόη έχει το λόγο. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για όλες τις πληροφορίες που μας έδωσε. Να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους. Έχω μια ερώτηση να κάνω. Θα ήθελα κυρίως να επιστήσω την προσοχή σας στο εξής. Υφίσταται μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δάση ή καλύτερα. Πολύ συχνά βλέπουμε ότι πρέπει να καταλάβουμε αν μια αποδάσωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία γίνεται για συγκεκριμένου οικονομικού ή βιομηχανικού λόγου, πραγματικά δικαιολογείται. Πώ μπορούμε δηλαδή να βοηθήσουμε κάποιε κοινότητε οι οποίε θέλουν να αναδασώσουν κάποιε περιοχές. Πώς μπορούμε λοιπόν να βοηθήσουμε τις εθνικές τοπικές αρχές, δημόσιες αρχές, να έχουν ένα καλύτερο συντονισμό με τους ιδιοκτήτες δασικών εκτάσεων προκειμένου να υπάρχει μια καλύτερη βιώσιμη διαχείριση των δασών. Θα μπορούσαμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να έχουμε help desks, κάποια κέντρα παροχής βοήθειας προς τους ανθρώπους αυτούς. Πρόεδρος, ο κύριος Ντόρφμαν έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πολλά ήδη υπόθηκαν σήμερα για την διαχείριση των ε, δασών. Έχουμε ακούσει διαφορετικές περιπτώσεις ε, για διαφορετικές ε, περιοχές. Σε ορισμένες περιοχές τα δάση προστατεύονται, σε ορισμένες χρήζουν προστασίας. Έχω να πω το εξής. Από ό,τι καταλαβαίνω, η προστασία του περιβάλλοντος και η οικονομική εκμετάλλευση βρίσκονται σε τη διαστολή αυτή τη στιγμή. Το αντίθετο θα έπρεπε να συμβαίνει. Εάν το δάσος δεν χρησιμοποιείται, παραμένει ένα κλειστό οικοσύστημα. Δεν παράγεται καινούρια ξυλία, δεν ε, δεσμεύεται περισσότερο διοξίδιο του άνθρακα εφόσον δεν υπάρχει καινούρια ξυλία. Το αντίθετο ε, με την ε, χρήση, την βιώσιμη χρήση των δασών. Μπορούμε έτσι να κάνουμε πολλά για το κλίμα Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε επίσης ε, τα δάση και για οικονομικούς ε, σκοπούς ε, για να εξοικονομήσουμε πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Η χρήση λοιπόν των δασών είναι πάρα πολύ σημαντική οικονομικά για πολλούς φορείς. Χρειάζεται όμως ε, αηφόρος χρήση και συνετή χρήση των δασών. Εσείς τι έχετε να πείτε γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπούντα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε, σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε εδώ ξανά. Θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή σε μια ιδιαίτερη περίπτωση που συμβαίνει στη Ρουμανία και σχετίζεται με την ε, δασοπονία. Η Δυνατότητα δηλαδή να φυτευτούν δάση σε οπορώνες ή σε περιοχές που δεν είναι πλέον καλλιεργήσιμες. Αυτό ε, είναι μια δυνατότητα. Η Ρουμανία όμως είναι δεσμευμένη να διατηρήσει ε, τις ε, περιοχές αυτές ανέπαφες μέχρι το 2016. Πρέπει λοιπόν από τη μία να Θα ήθελα επίσης να πω ότι χρειάζεται να γίνει μια διεξοτική συζήτηση. Χρειαζόμαστε ένα διαφορετικό πρόγραμμα από το πακέτο στήριξης, διότι αυτό το πακέτο στήριξης είναι ε, γελίο σε σχέση με τα ποσά που πραγματικά χρειάζονται για να στηριχθεί ο τομέας των ε, γαλακτοπαραγωγών. Πρέπει να αντισταθούμε και να αντιδράσουμε σε αυτήν ε, την ε, αυτόν τον πόλεμο που γίνεται αυτή τη στιγμή προς τους παραγωγούς γάλακτος. Σας ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, τελειώσαμε τώρα. Με τον κύκλο θα δώσω τώρα τον λόγο στον Επίτροπο και θα ήθελα να τον παρακαλέσω να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ε, να απαντήσω πρώτα σε αυτά τα οποία δεν είναι δασικά. Τα είπαμε τα είπαμε και στην Ολομέλεια του Σεπτεμβρίου. 52 άτομα, κυρίως από αυτή την επιτροπή, μίλησαν για το γάλα. Ξέρετε τι έχουμε πληρώσει σε άμεσες ενισχύσεις. Ξέρετε τι έχουμε ε, στην ε, συνδεδεμένη βοήθεια ε, και πώς έχουμε στηρίξει με τον τρόπο αυτό την ντόπια παραγωγή. Ξέρετε τι συμβαίνει ε, στη Γερμανία με το γάλα. Η τιμή είναι κάτω από την... Ε, ε, η τιμή στην οποία πωλείται το γάλα είναι χαμηλότερη από την τιμή που κοστίζει να παραχθεί και παρόλα αυτά συνεχίζουν την παραγωγή. Γιατί? Γιατί στηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βεβαίως τα στοιχεία είναι πάρα πολύ δύσκολα να τα πιστέψει κανείς, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Για το γάλα στα σχολεία, εμείς όντως θα δώσουμε παραπάνω κονδύλια. Θέλουμε μέχρι τα τέλη της χρονιάς να έχει κλείσει το θέμα αυτό, ε, έτσι ώστε να αναθεωρηθεί το πρόγραμμα αυτό και το έχουμε ήδη ανακοινώσει. Να σας πω καταρχήν πως δεν είμαι ανακριτής. Ούτε detective. Επίτροπος είμαι. Δεν μπορώ να κάνω στην DG Agri. Είναι θέμα αρχών και νομίζω ότι εκεί έπρεπε να φάει ο φάκελος και πολύ σωστά κάνατε. Νομίζω ότι η Γκάρντα, δηλαδή η αστυνομία στην Ιρλανδία, είναι η κατάλληλη για να το ερευνήσουν. Για τα δασοκομικά θέματα να σας πω πως τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης στην Ιρλανδία έχουν αυξήσει το δασικά εδάφη στο 18%. Άρα λοιπόν θα έχουμε μεγάλη ζήτηση ε, και για τα προϊόντα βιομάζας και ε, για τα υπόλοιπα δασικά προϊόντα πολλοί πορεί έχουν ε, διατεθεί μέσω των προγραμμάτων ε, επιστήμης, έρευνας, τεχνολογίας και εδώ θα συμπεριλάβουμε και άλλους κλάδους της βιοοικονομίας πιο γενικά. Ελπίζω λοιπόν πως σύντομα ε, οι δείκτες που θα παρουσιάσουμε θα αποδείξουν πόσο καλό τι είμαστε και το πόσο θέλουμε η χρήση γης να συμπεριλάβει και τη δασοκομεία σε περιοχές για παράδειγμα όπως στη Σλοβενία που μίλησε ο κύριος Μπόκοβιτς για το 60% ε, που, της γης που καλύπτεται από δάση και που θέλει να γνωρίζει καλύτερα πώς μπορεί να προσελκύσει θέσεις εργασία στην περιοχή χρησιμοποιώντας αυτή τη στρατηγική. Τώρα, η, η, η δάση Ήρθαμε σε επαφή με τη σχετική ομάδα εργασίας για το πολιτέ ε, και θα ε, συμμετέχουν και αυτοί στην εφαρμογή. Και ξέρετε πως πρόεδρος της ομάδας είναι ένας ιδιοκτήτης δάσους. Ελπίζω αυτό λοιπόν ε, να καθησυχάζει τον ιδιωτικό κλάδο. Δεν σας έχουμε αγνοήσει. Κύριε Μπούτα, τις λεπτομέρειες να μου τις στείλετε, γιατί είναι πολύ τεχνικά τα ζητήματα και θα τα ψάξω. Ο κύριος Άγνιο αναφέρθηκε στο γεγονός ότι δεν υπάρχει κοινή δασική πολιτική όπως δεν υπάρχει ΚΑΠ. Όμως έχουμε κοινή στρατηγική για τα δάση. Και γιατί πρέπει να παίζουμε αυτό το ρόλο. Γιατί έχουμε τα 7,2 δος δις από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Άρα λοιπόν πρέπει να προστατεύσουμε τα συμφέροντα του Ευρωπαίου φορολογούμενου. Αλλά βεβαίω εδώ ε, μιλάμε για το ρόλο του κράτους μελού στην εφαρμογή της πολιτικής δεν αναφέρεται στην ε, συνθήκη και δεν το προτείνουμε αλλά νομίζω ότι υπάρχει εδώ μια ευκαιρία να προσφέρουμε προστιθέμενη αξία θέσεις εργασίας στην Ήπεθρο ε, και να τα πάμε καλύτερα από ό,τι τα πάμε σήμερα. Και ξέρετε τι συμβαίνει στη Φιλανδία. Καλό είναι λοιπόν να έχουμε μεγάλες επενδύσεις εκεί για να έχουμε θέσεις εργασίας. Εκεί βέβαια είναι πιο εύκολο από ό,τι σε άλλες περιοχές. Δεν προτείνω λοιπόν εγώ κοινή δασική πολιτική με τον παραδοσιακό τρόπο που έχουμε την κοινή αγροτική πολιτική αλλά πρέπει εμεί να εξασφαλίσουμε πως τα χρήματα αυτά χρησιμοποιούνται με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο για να πετύχουμε τους στόχους μας λαμβάνοντας υπόψη πάντα την επικουρικότητα. Πάλο. Εμείς περιμένουμε την τελική εκδοχή και γι' αυτό ζητήσαμε τη γνώμη του ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αλλά το ξέρεις άλλωστε. Για να είμαστε σίγουροι πως τα θέματα τα οποία θίγουν οι ευρωβουλευτές λαμβάνονται δεόντως υπόψη. Και σου υποσχέθηκα πως θα σε ενημερώνω πάντα με το πώς πάει η εφαρμογή του πολίτους. Τώρα, πρώτες ύλες για τη βιοοικονομία. Έτσι μπορούμε να κατακτήσουμε νέες αγορές, να διαφοροποιήσουμε αγορές, αλλά βέβαια βιώσιμη διαχείριση δασών είναι μια πρόκληση και η ισορροπία μεταξύ συμφερόντων επίσης. Όπως επίσης και ο σεβασμός βιωσιμότητας και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε στενή συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς και τα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν τα σημεία αυτά. Φετηρία και βάση της εργασίας μας είναι και αυτό το έχουμε α, αναλύσει υπό τους τρέχοντες δείκτες είναι το Forest Europe και το πώς αυτά εφαρμόστηκαν. Έχουμε μια έκθεση της ομάδας εργασίας στην οποία συμμετείχαν πάρα πολλοί ε, εμπειρογνώμονες και εμπλεκόμενοι φορείς ε, που εγκρίθηκε μόλις από τη Μόνιμη Επιτροπή για τα δάση. Η νέα πολιτική βιομάζας θα πρέπει να συμπεριλάβει την βιώσιμη διαχείριση δασών που θα φιδεγαμίζεται με την πολιτική μας και να δει ποιες είναι οι έμεσες συνέπειες χρήσης γης, όπως είπατε και εσείς, πώς επηρεάζει ε, η αλλαγή του κλίματος. Αυτή τη στιγμή περνάμε τη φάση αξιολόγησης. Πρόσφατα ε, ατύπως συναντηθήκαμε στη Ρία και με τους Υπουργούς ε, Ενέργειας για να δούμε ποιες είναι οι προκλήσεις και να εντοπίσουμε τους κινδύνους που θα προκύψουν από τις ΑΠΕ ε, και... Ε, να βρούμε μια λύση η οποία θα είναι ευνοϊκή για όλους. Εγώ είμαι σε ε, επαφή με τον Επίτροπο που ε, ασχολείται με τα θέματα κλιματικής αλλαγής. Δεν έχουμε καταλήξει ε, σε συμπεράσματα, αλλά σίγουρα η δασοκομεία θα είναι βασικός παράγοντας και ο τρόπος που επηρεάζουν τα δασικά προϊόντα θα χαράξουν σε μεγάλο βαθμό τη στρατηγική μας. ΑΠΕ, βιομάζα, μέχρι στα πλαίσια της στρατηγικής για το 2020 η χρήση της βιομάζας ε, λαμβάνεται ε, όλο και περισσότερο υπόψη και στην εφαρμογή της στρατηγικής ε, τα κράτη-μέλη θα λάβουν τις προτάσεις που θα κάνουμε εμείς στην αναθεώρηση του 2016 για παράδειγμα βιομάζα στις συγκοινωνίες, βιομάζα στην θέρμανση και στην παραγωγή ενέργειας. Μπορούμε να δούμε τη βιομάζα στα πλαίσια του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης σε όλα τα κράτη-μέλη με βιώσιμη ε, παραγωγή ε, δασικής ε, προέλευσης βιομάζας έτσι ώστε να έχουμε την κατάλληλη και βιώσιμη προώθηση και εμπορία. Επίσης, νέες αλυσίδες παραγωγής. Για παράδειγμα, προώθηση και μάρκετινγκ της βιομάζας. Τα κράτη-μέλη θα αποφασίσουν ποια μέτρα θα συμπεριλάβουν ε, στην αγροτική ανάπτυξη. 3,3 ε, δις πάντως έχουν ε, περιχαρακωθεί, οπότε εμείς θα δούμε πώς θα εφαρμοστεί και πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα τμήμα αυτών των κονδυλίων και για την πρόθεση βιομάζας. Τελικά, το αυτό που μπορώ να πω είναι οι αγορές ξύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ακολουθούν τους κανόνες της προσφοράς και της ζήτησης. Εμείς απλώς θα οριοθετήσουμε τις αγορές αυτές έτσι ώστε κάποια στοιχεία όπως οι φυτογειονομικές ε, διατάξεις ε, και κάποια άλλα θέματα βιωσιμότητας να γίνουν σεβαστά. Πρώτες ύλες πρέπει να χρησιμοποιούνται με τον τρόπο που προσθέτει αξία που ε, χρησιμοποιείται για όλες τις ανάγκες που καλύπτει το ξύλο και οι πόροι να κατανέμονται με ισόρροπο τρόπο έτσι ώστε η αγορά ξύλου να λειτουργεί σωστά. Αυτό πρέπει να αξιολογηθεί και να λάβει υπόψη και, τις, ε, ε, και τη δομή των δασών αλλά και των αγορών δασικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πυρκαγιές δάσους, αυτό το βλέπουμε στο ΕΤΠΑ για το 2014-2020, φυσικές καταστροφές στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, για παράδειγμα ανώτος της Γαλλίας, πρόσφατα όσα συνέβησαν, το, το πρόγραμμα αγροτική ανάπτυξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί έτσι ώστε να έχουμε κάποια μέτρα αναδάσωσης για παράδειγμα ή ανοικοδόμηση ή ανασυγκρότηση όταν έχουμε τέτοιου είδου φυσικές καταστροφές και βεβαίω θα ήθελα να εκφράσω και τα συλληπιτήριά μου στι οικογένειε των θυμάτων. Μέσω του συστήματος ε, ενημέρωσης για δασικές πυρκαγιές και τον χάρτη έγκαιρης προειδοποίησης έχουμε μια βάση δεδομένων με τους κινδύνους και είμαστε σε στενή επαφή με τα κράτη-μέλη και με την σχετική ομάδα εμπειρογνωμόνων. Έχουμε επίσης τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας για την πρόληψη καταστροφών που απαιτεί από τα κράτη-μέλη να κάνουν αξιολόγηση κινδύνων σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και να μας, ε, μοιραστούν μαζί μας το δυναμικό που έχουν ε, για τη διαχείριση των κινδύνων αυτών. Στην περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 προβλέπουμε κονδύλια προκειμένου να γίνεται μια σωστή χρήση όλων αυτών των μέτρων ε, πυρασφάλειας. Όλα αυτά τα μέτρα προστασίας των δασών από τις ε, πυρκαγιές αποτελούν ε, αρμοδιότητα των κρατών μελών, αλλά πρέπει να υπάρχει συντονισμός ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Η νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δάση επίσης δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα προϊόντα του δάσους, τα οποία δεν αποτελούν ξύλια. Πέρα από την ξύλια δηλαδή και αυτά τα προϊόντα μπορούν να συμβάλλουν πάρα πολύ στην ε, ανάπτυξη της υπαίθρου. Δίνονται λοιπόν οι απαραίτητες δυνατότητες προκειμένου να προωθήσουμε όλους αυτούς τους παρεμφερείς εκτός ξυλίας. Μας ενδιαφέρουν επίσης όλες οι σχετικές οικοσυστημικές υπηρεσίες που δεν σχετίζονται με την ξυλία και πώς αυτές θα μπορούσαν να συμβάλλουν περισσότερο στις αγροτικές περιοχές. Στα πλαίσια της στρατηγικής αυτής θέλουμε να μειώσουμε της ε, τάσης υπερβολικής κατανάλωση σε παγκόσμιο επίπεδο και να προωθήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο την ε, βιώσιμη διαχείριση των δασών και να πετύχουμε και την κατάλληλη συνεργασία όχι μόνο μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσπαθούμε λοιπόν να μειώσουμε με τους διεθνείς εταίρους μας τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα που προκύπτουν από την, αποδάθ, από την αποδάσωση και θέλουμε να καταφέρουμε να εντάξουμε συγκεκριμένους δείκτες στη διαδικασία Ρίο Κύριε Πρόεδρε, ενδεχομένως να μην κάλυψα τα πάντα, πάντως σε κάθε περίπτωση μπορώ να σας αποστείλω και περισσότερες απαντήσεις στα ερωτήματα τα οποία μου θέσατε. Αν έχετε θίξει τεχνικά ζητήματα θα ήθελα να έχω τη δυνατότητα να σας απαντήσω σε αυτά σας Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Συντοπίμε όλοι ότι τα δάση αποτελούν έναν χώρο στον οποίο συμβάλλουν ή τον οποίο επηρεάζουν πολλές πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι μόνο η γεωργία και η ανάπτυξη πέθρου, είναι και η πολιτική μας για την ενέργεια, την κλιματική αλλαγή που επηρεάζει τον τομέα των δασών. Απαιτείται λοιπόν συντονισμός ανάμεσα στις διάφορες πολιτικές. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δάση. Γνωρίζουμε επίσης κύριε Επίτροπε ότι τα δάση αποτελούν αρμοδιότητα εθνική, σίγουρα. Ωστόσο, συνειδητοποιούμε επίσης ότι ε, υφίστανται αυτή τη στιγμή κάποιες επιτροπές, κάποιοι οργανισμοί, οι οποίοι ε, προσπαθούν να διασφαλίσουν ότι υπάρχει μια συντονισμένη ευρωπαϊκή διεθνής δράση. Πολλές συνδιασκέψεις ε, λαμβάνουν χώρα αυτή τη στιγμή, διοργανώνονται από διάφορους φορείς παντού στην Ευρώπη και υποστηρίζονται από διάφορες επιτροπές και στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέλουμε λοιπόν μια τέτοια ενσωμάτωση. Χρειαζόμαστε επίσης και την κατάλληλη χρηματοδότηση. Χωρίς χρηματοδότηση δεν μπορούμε να πετύχουμε τίποτα. Κύριε Επίτροπε, για άλλη μια φορά σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοδομητική αυτή συζήτηση που έλαβε χώρα. Υπάρχουν κάποια ζητήματα τα, πιέζουν, τα οποία πιέζουν πάρα πολύ, όπως για παράδειγμα η κρίση στον γαλακτοκομικό τομέα. Κύριε Επίτροπε, φαντάζομαι ότι δεν σας κάνει εντύπωση το ότι ε, θίξαμε το ζήτημα αυτό, ερχόμαστε όλοι σε επαφή με, τις, με τους εκπροσώπους των εκλογικών μας περιφερειών. Όλα αυτά αποτελούν μέρος της καθημερινής μας ζωής. Αυτό δεν σημαίνει ότι ξεχνάμε και τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δάση. Άλλωστε η συγγήτριά μας η κυρία Κέστιγκερ αναφέρθηκε πολύ καλά στο ζήτημα αυτό. Για άλλη μια φορά κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμβολή σας. Θα συναντηθούμε πάλι την Δευτέρα στις 3 το μεσημέρι. Και στη συνέχεια την Τρίτη θα ξεκινήσουμε την, μια πολύ δύσκολη ψηφοφορία στις 9 το πρωί θα ψηφίσουμε την έκθεση Hoistling και το απόγευμα θα συνεχίσουμε πάλι τη συνεδρίασή μας, το απόγευμα της Τρίτης δηλαδή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν για την ε, συμμετοχή σας και μην ξεχνάμε ότι έχουμε και πολλά άλλα σημαντικά γεγονότα στην Σύνοδο Λομέλειας αυτή την εβδομάδα εδώ στο Στρασβούργο. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ σε όλους και για άλλη μια φορά επίτροπες, ευχαριστούμε πολύ.